κυρία Πλινκοβιτέ, θα διενεργήσει τις πληροφορίες εκ μέρους μου. Ε, κοινή συνεδρίαση ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ε, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπλέμψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Είμαστε έτοιμοι. Καλωσορίζω την κυρία Πλάνκοβιτσίουτε από την Επιτροπή Γυναικοματογυναικών. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Συμβαστική παρθμόν 1. Για τα μέλη της Επιτροπής ε, ΦΑΜ όλα γίνονται ηλεκτρονικά, επειδή δεν το ξέρετε. Εντάξει. Δεν σηκώνουμε χέρια. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Όχι. Ωραία. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή Γυναικών χωρίς την κάρτα του. Στη Λίμπε όλοι έχουμε κάρτες μαζί μας βέβαια. Ή μιλήστε τώρα ή σιωπήστε για πάντα. Ε, ωραία. Συμβαστική παρθυμόν 1. Έναρξη. λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική παρθμό 2. Λήξη. Εγκρίνεται. Σε συμβαστική 2α. Έναρξη. Ψήφισαν όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Τροπολογία 203. Προσθήκη. Πολύ 203. Έναρξη. Είναι προσθήκη. Μόνο την προσθήκη ε, ψηφίζουμε. Μόνο την προσθήκη. Ψηφίσαμε ήδη την προσθήκη. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 200... Ε, συγγνώμη, τροπολογία 204, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 213 εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 5 έναρξη. λήξη. Εγκρίνεται συμβαστική παριθμόν 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται συμβαστική παριθμόν 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται συμβαστική παριθμόν 8. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 9. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 9α. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 252. Έναρξη. Απορρίπτεται. 253-251 δεν μπορούμε να τις πάρουμε όλοι μαζί. 253 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 2.54 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 2.51 έναρξη. Φαντάζομαι και αυτή θα απορριφθεί. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμόν 11. Έναρξη. έναρξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 12. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 13. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 14. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 283. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 284. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 15. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 291, ε, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Συμβαστική 16, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 298, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 302. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 303 και 307 είναι ταυτόσιμες. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 305 και 306 πάλι ταυτόσιμες. 26 απορρίπτονται. Τροπολογία 309 και 312 ταυτόσιμες έναρξη. Δεξί. Απορρίπτονται. Τροπολογία 310 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτονται. 311 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 313 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 314 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 3.15. Λήξη. Εγκρίνεται. 2.48. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δύο, ε, συγγνώμη, 3.16. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 3.17 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε όλοι μαζί το blog α, για τις αναφορές και την ε, αιτιολογική έκθεση. Λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο μπλοκ, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμών 3. Έναρξη. Λήξη. Έγκρινεται. Συμβαστική 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστη... Συγγνώμη, τροπολογία 66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Κατά τμήματα, το τμήμα του ΕΛΚ, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 73. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 100. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 76. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 98. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαντική τέσσερα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. δύο. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη. Απορρίπτεται. 103. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 104. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 117. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Συμβαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 122. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ταυτόσιμες 120. 143, 183. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 133. Άρχεται. Πέρας. 134. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 136. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 137. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 138. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 140 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαντική εννέα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 148. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 156. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 156. Ωραία, εγκρίνεται. 157. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 158. Άρχεται. Δική σου μου το σωστά. 158. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 168. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 170. Άρχεται. Απορρίπτεται. 191. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 192. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 173. Άρχεται. Πέρας. Κύριε Άγγελ, κύριε Λέναρτς, μην περνάτε τόσο ωραία. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Λυπάμαι για τα μέλη του ΕΛΚ. Λοιπόν, 174. Άρχεται. 174. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. 175. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 181. Άρχεται. Πέρας. Πριν την τελική ψηφορία Ζητώ συγγνώμη και από τον Συμπρόεδρο, δεν αναφέραμε τους συζητητές. Ευχαριστώ την Άννα Μαρία Κορέτσα Μπίρτ και την κυρία Μπονεφόη, συνεισυγήτρια σε αυτήν την έκθεση. Θέλω να τις ε, ευχαριστήσω και να τις χαρώ. Ναι, το κάνω τώρα, γιατί ξέρω ότι με το που θα έχουμε την τελική ψηφοφορία όλοι θα φύγετε. Είμαι βέβαιος βέβαια ότι θα είστε τόσο ευγενείς που θα μείνετε για τα κατακλητικά μου σχόλια. Τέλος πάντων, με ονομαστική κλίση, όπως έχει τροποποιηθεί το κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Και τώρα μπορείτε να αποχωρήσετε. Πέρας. Εγκρίνεται 58 υπέρ 12 κατά 4 εποχές. Συγχαρητήρια στις εισηγήτριες. Thank you very much. Thank you, colleagues. Madam Saborska, do you want to say a quick word, please? Go ahead. Κυρία Σαμπόσκα, θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει του κανόνα 52α. Θα ήθελα να υποβάλω ε, τη θέση μου για αυτή την ψηφοφορία. Επίσης, Θα τη στείλω και γραπτός στη γραμματεία. Ευχαριστούμε. Κύριε Τζούρεκ, και εσείς το ίδιο. Ναι, μάλιστα. Και εγώ θα υποβάλω γραπτά σχόλια. Ωραία, ευχαριστούμε. Thank you. Thank you, colleagues. Have a good summer if I don't see some of you.